Ευχαριστώ πολύ. Ε, πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την ε, έκθεση Σάντσε Σμιτ, Ευρωπαϊκή Τομή του Πολιτισμού και της Δημιουργίας ως πηγές οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Merci, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο τομέα του πολιτισμού και τη δημιουργία ενισχύει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλό αυτό ο τίτλο. και αυτό ακριβώ είναι και ο στόχο τη έκθεσής μου, να επιτρέψουμε στο δυναμικό του πολιτισμού και τη δημιουργία να αναπτυχθεί. Ο στόχο είναι σαφή. Τώρα που βρισκόμαστε σε κρίση πρέπει να προσφέρουμε συγκεκριμένε λύσει για να ενισχύσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη. Όμω η τομεί του πολιτισμού και τη δημιουργία δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη παρόλα αυτά προχωρούν παρά την κρίση, αντιστέκονται στην κρίση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και εμπίπτουν κάλλιστα στη στρατηγική του 2020 για μια ευφυή βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία να συμμετέχουν όλοι. Προωθεί την καινοτομία, την δημιουργικότητα, την ε, κατάρτιση που είναι έτσι πιο ανοιχτή στον κόσμο εφόσον λαμβάνει υπόψη τον πολιτισμό και τη δημιουργία. Τα 20 τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με εκθετικό τρόπο. Πάνω από 8 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ο τζίρος και πάνω από 8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Έχει τεράστιο δυναμικό ο τομέας αυτός τώρα μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να πιστούν να επενδύσουν στον πολιτισμό και την δημιουργία, γιατί τα ενδυνάμει κέρδη είναι τεράστια. Υπάρχουν περιφερειακά φόρα, υπάρχει το ε, περιφερειακό ταμείο, υπάρχει το φεστιβάλ της, ε, των κανόνων, της Αβινιών κλπ που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις περιφέρειες όπου βρίσκονται και στις κοινωνίες που ζουν σε αυτές. Τα ευρωπαϊκά ταμεία λοιπόν πρέπει να στηρίξουν τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και να αναγνωρίσουν τα οικονομικά εφέλη από αυτούς. Τα οικονομικά ωφέλη είναι τεράστια. Συνεισφέρουμε επίσης την πολιτισμική πολυμορφία είναι αναγκαίο να υπάρξει νέος δυναμισμός από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να ενισχύσει την ανάπτυξη των τομέων αυτών με ρύθμιση για την τον ανταγωνισμό, για φορολογικά στοιχεία, για την κατάρτιση των δημιουργών, για το ψηφιακό χαρακτήρα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για τον υποτιτλισμό, για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, της πνευματικής ιδιοκτησίας, ένα νομικό πλαίσιο που να είναι ελκυστικό, εκδόσεις. Όλα αυτά είναι τομείς δραστηριότητας που μπορούν να συνεισφέρουν στον πλουραλισμό των μέσων και την πολιτισμική πολυμορφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει λοιπόν να στηρίξει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, να ενισχύσει την, καινοτομία, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και να επιτρέψει την κατάρτιση, την ανοιχτή στον κόσμο. Πρόκειται για τεράστια προστιθέμενη αξία με κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία σε όλες μας τις χώρες. Η τεχνολογία επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη που μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την καινοτομία με επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη είτε πρόκειται για τοπικό είτε πρόκειται για περιφερειακό επίπεδο, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης πολύ περισσότερες από ότι όλοι οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν μοχλός ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργίας για την ανάπτυξη των οικονομιών μας, με θέσεις απασχόλησης. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά χάρη στους τομείς αυτούς μπορεί να αντισταθεί και να ε, έχει κέρδη από την παγκοσμιοποίηση μέσω της δημιουργίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιωτερότητες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος είναι ο κύριος Λόπες Ιστουγκάιτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Μαρή Τερέ Σάντσε Σμιθ θέλω να υπογραμμίσω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους νέους δημιουργούς πάνω απ' όλα. Ο πολιτισμός αποτελεί στοιχείο κοινωνικής συνοχής. Με την τεράστια ανεργία των νέων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ ο πολιτισμός να αποτελέσει μια ευκαιρία για τους νέους δημιουργούς. Όχι πολιτισμό επιδοτούμενο, όχι, αντίθετα να μπορούν οι δημιουργοί να φτιάξουν τις δικές τους μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ευκαιρίες για άλλους. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, την ε, πολιτισμική εξαίρεση. Ελπίζω να βοηθήσει περισσότερο. Και όπως ε, ακούσαμε πριν, οι τομείς αυτής ενισχύουν και το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό πέρα από το περιφερειακό και το τοπικό. Ευχαριστώ πολύ. the next speaker is Επόμενη ομιλητή η κυρία Γκρίσμπεκ. Yeah, there is a blue card. Δέχεστε την γαλάζια κάρτα. Mr. Uh, θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Ροκάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής ε, Πολιτισμού θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεισφορά της στην ε, πολύ σημαντική αυτή συζήτηση. Ε, ελέγχθη ότι το μέσο του πολιτισμού μπορεί να βοηθήσει για να βγούμε από την κρίση ε, και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και συμφωνώ με αυτό αλλά διαβάζοντας την έκθεση ε, με κάποια απογοήτευση διαπιστώνω ότι υπάρχει ένας βαθμός προστατευτισμού Ε, υπάρχει εντύπωση ότι μπορούμε να ε, προστατεύσουμε τη δημιουργικότητα με ε, μέτρα τα οποία δεν θα επιτρέψουν στα αμερικανικά προϊόντα να πλήξουν την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα. Πιστεύω ότι αυτό εις βάρος μας θα είναι μάλλον παρά εις όφελός μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή ελεύθερη αγορά στο μέτρο του δυνατού. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός θα επιβιώσει και είμαι βέβαιος ότι και η Γαλλία και η Δανία και όλες οι άλλες χώρες θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα στον ανταγωνισμό με τους Αμερικανούς στον πολιτιστικό τομέα και πιστεύω από πλευρά τη Δανική αντιπροσωπεία ότι δεν μπορούμε να βάλουμε αυτή την πολιτιστική εξαίρεση μέσα στις διαπραγματεύσεις ε, για το ελεύθερο εμπόριο. Είναι πολλά αυτά τα οποία διακυβεύονται με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σπάσκα. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις για την πράσινη βίβλο, για τις δημιουργικές πηγές της οικονομίας είναι στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να πούμε ότι παρά το ότι αυτό ήταν γνωστό η Επιτροπή αυτή τη στιγμή η Κομισιόν μας δίνει και νέες οθήσεις αν και δεν τα έχει λάβει όλα υπόψη της όσα θα έπρεπε ας πούμε ανθρώπους που αρχίζουν μία μικρή επιχείρησή τους στον καράζ τους είναι γνωστό ότι σήμερα έχουν φτάσει να καθορίζουν τα πρότυπα της επικοινωνίας παγκόσμια όπως η Apple και η ίδια και η Microsoft με την Google είναι γνωστό τι επιτυχία και τι ρόλο παίζουν. Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία στην οικονομία αλλά πρέπει να βοηθήσουμε την εφαρμογή μέτρων προώθησης της. Να προωθηθεί η δημιουργικότητα δηλαδή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα λάβει το λόγο η Επίτροπος Ρέντινγκ. Κύριε Πρόεδρε, Ξέρετε, κύριε βουλευτέ, η Κομισιόν καλωσορίζει την προσέγγιση για την ολοκληρωμένη υποστήριξη προς ε, του τομεί του πολιτισμού και τη δημιουργία. Ε, νομίζω ότι έχουμε μια κοινή πεποίθηση. Αυτή η τομή είναι μεταξύ των πλέον υποσχόμενων στην Ευρώπη σήμερα. Μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στη στρατηγική δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη και γι' αυτό η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ε, πολλαπλέ στρατηγικέ πολλαπλών στρωμάτων για να προωθήσουν ε, το δυναμικό του πολιτισμού και τη δημιουργία και να θέσουν αυτή τη στρατηγική υψηλά στην ημερήσια διάταξή τους. Η στρατηγική που προτείνεται από την ανακοίνωση και το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημιουργική Ευρώπη είναι σημαντικά οχήματα για αυτή τη φιλοδοξία. Η Κομισιόν με ικανοποίηση συμμετέχει ότι η έκθεση της κυρίας Σάντσες Μη θα αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Παραδείγματος χάρη το να αναπτυχθούν δημιουργικές δεξιότητες σε ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, προκλήσεις ε, της παγκοσμιοποίησης ε, και της νέας ψηφιακής εποχής, της ψηφιοποίησης και η δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Η Κομισιόν ε, έχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα, αλλά επίσης ε, έχει καταρτήσει και μια βραχυπρόθεσμη πρακτική στρατηγική με συγκεκριμένους άξονες ε, που θα υλοποιηθεί με συντονισμένες δράσεις τα επόμενα έτη η νέα γενιά της ε, χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2014-2020 θα δώσει πολλές ευκαιρίες για τους τομείς της δημιουργίας. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα βοηθήσει τους καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες και τις οργανώσεις να εργαστούν διασυνοριακά και να απευθυνθούν σε ένα ευρύ κοινό. Είναι δυνατό η πολιτιστική κοινότητα και η τοπική αυτοδίκηση να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το περισσότερο κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν καλωσορίζει τη συνεισφορά που μπορεί να κάνουν αυτοί οι τομείς για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη. Ευχαριστούμε κυρία Ρέντιν, κυρίες και κύριοι. Έληξε αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12. 12. Eh, Επόμενο θέμα της στην ημερήσια διάταξη είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Δήλωση της Επιτροπής. Όπως βλέπετε τώρα κάθε